Υποδεχόμαστε την Βία Ντακέλ που είναι συνάδελφος ε, βουλευτής στο Ιρακινό Κοινοβούλιο. Κανείς δεν θα ξεχάσει ποτέ την συγκινητική της ε, ομιλία την οποία έκανε το περασμένο Αύγουστο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου της χώρας του που ζητούσε παρέμβαση για την απελευθέρωση των γυναικών της ε, κοινότητας των γυναικών Γεζιντή που έχουν συλληφθεί από το Ισλαμικό κράτος όπως αυτό αποκαλείται συνοδεύεται από μία αποστολή ε, ε, γυναικών Γεζιντή, την κυρία Εσβάτ ε, Ασάν, την κυρία Οτμάν, το κύριο Κορσέτ Οτμάν Γιουσίφ εμείς όλοι μας σας τιμούμε σας τιμούμε για το θάρρος σας και σας ε, διαβεβαιούμε για την απόλυτη μας υποστήριξη στον αγώνα και στο δικαίωμα του λαού Γεζιντή να ζήσει με αξιοπρέπεια και να ασκεί ελεύθερα την θρησκεία του. Καλωσορίσατε στο Στρασβούργο, καλωσορίσατε στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην αίθουσα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας.